Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Όπως λέει και ο πρόεδρος Ντεάν, πέρασε το ακαδημαϊκό τέταρτο και ο εισηγητής μας μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Υπάρχουν όμως δύο ενοχλητικοί οι οποίοι την εμποδίζουν να συγκεντρωθεί. Σήμερα το πρωί πήγαμε πολύ γρήγορα και ελπίζω ότι με την ίδια ταχύτητα θα προχωρήσουμε και σήμερα το απόγευμα όπου θα ψηφίσουμε τις ε, ε, τροπολογίες για τη Γαρία 3α και 3β. Δεν μπορούμε ακόμη να ψηφίσουμε την κατηγορία 4 διότι δεν, έχουμε, δεν ξέρουμε ακόμη πόσο θα προχωρήσουμε άρα αυτό θα απασχολήσει τους συντονιστές ε, οι οποίοι θα συνεδριάσουν μετά και αύριο το πρωί θα ψηφίσουμε την κατηγορία 4 και τις πυρλωτικές ε, δράσεις καθώς ε, και τη γραμμή ίτερ και ορισμένες άλλες επί των οποίων ενδέχεται να μην έχουμε βρει μία ικανοποιητική λύση εχθές και σήμερα. Λοιπόν, Εάν τελειώσουμε λοιπόν γρήγορα θα μπορέσουμε ε, να έχουμε τους συντονιστές με διερμηνές και να σας αποδεσμεύσουμε για να κάνετε πιο ευχάριστα πράγματα από το να ψηφίζετε. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το 3α αμέσως. Στο αγγλικό κείμενο είμαστε σελίδα 106 η γενική επικεφαλίδα στο 3α είναι Citizenship, Freedom, Security and Justice. Δηλαδή ε, οι πολίτες, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Και ξεκινάμε με την τροπολογία 4673, αλλά μου λένε ότι επικαλύπτεται. Όχι, λοιπόν... Ε, ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 4673. Ο κύριο ε, Χάρτουν και η κυρία Αντρέσεν. Απορρίπτεται. Δεν είναι η συνήθις ε, τροπολογία Ερεν Χάουζερ, αλλά αυτή η απόφαση ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Το επόμενο έχει καλυφθεί, πρέπει όμως να ψηφίσουμε την 196. Η συγγήτρια. Για τη 18.04.03 ουσιαστικά είχαμε ψηφίσει την αποκατάσταση του προσχεδίου χθες, αλλά υπάρχει αίτημα για ξεχωριστή ψηφοφορία της ομάδας Άλντε νομίζω είναι το αίτημα. Όχι των σοσιαλιστών είναι. Για να ψηφίσουμε τα 50.000 που λείπουν ακόμα. Γιατί είχαμε ψηφίσει για την οριζόντιο χθε και ήταν 50.000 να προσθεθούν. Είμαι κατά όμως αυτής της αύξησης εγώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελικά, τι αριθμό πρέπει να τοποθετήσουμε εδώ, σε αυτή την τροπολογία. Η κυρία Γιάνσεν. Πρόεδρε, ειλικρινά, αν ψηφίσαμε ένα κονδύλιο, ψηφίσαμε ένα πακέτο μέτρων και θα πρέπει να καλύπτεται αυτό. Δεν ξέρω πώς ψηφίσαμε ένα πακέτο και αυτό εξαιρείται από το πακέτο και το ξαναψηφίζουμε. Ψηφίσαμε ένα ολόκληρο πακέτο ως μέτρα. Okay. Donc je ne soumets pas au vote οπότε δεν θα ψηφιστεί. Λοιπόν, προχωράμε. Το 4672 καλύφθηκε, ενώ η 197 έχει καλυφθεί και αυτή. Ωραία. Βρισκόμαστε λοιπόν στην 106 αγγλικού κειμένου και προχωράμε στην 107 αγγλικού κειμένου. Όλα έχουν καλυφθεί. ακόμη και η τροπολογία 200 μου λέγεται. Θα με διορθώσετε εάν κάνω λάθος και φτάνουμε στη σελίδα 108. Το 4677 του κυρίου Έρεν Χάουζερ. είναι δηλαδή ε, μία καταρχήν, ε, ποιος είναι υπέρ, καταρχήν ε, μείωση κατά 10 ή 15% θα τη βρούμε και στη συνέχεια. Οπότε αυτή η πλειοψηφία θα ισχύσει με τις ε, ίδιες, ε, τις ίδιες ε, τροπολογίες Ερενχάουζερ όπως έγινε και στα προηγούμενα κεφάλαια και για τους πράσινους για τη γεωργία. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με τις δύο επόμενες τροπολογίες Χάουζερ. Ε, έχουμε την τροπολογία χάρτου 4159 και το ψηφίζουμε γιατί είναι μια νέα κατηγορία. Ποιο είναι υπέρ. Υποθέτω ότι ο κύριος Χάρτουγκ είναι υπέρ και η κυρία Αντρέσεν ποιοι είναι κατά. Και αποχές. Λοιπόν, και εδώ θα ισχύσει το ίδιο καθεστώς. Σε τέτοιες τροπολογίες του κυρίου Χάρτον θα θεωρήσουμε ότι αυτή η ψηφοφορία καλύπτει τις περιπτώσεις. Το 630, η συγγήτρια είναι κατά. Έχει αποσυρθεί. Με συγχωρείτε, εγώ έκανα λάθος. 43-59 καλύπτεται επίσης, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε το 205. Ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη ε, καλύπτεται και ερχόμαστε στη 201. Ποιος είναι υπέρ, η εισηγήτρια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 524. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. ηλεκτρονική ψηφοφορία διότι αντιλαμβάνουμε ότι δεν συμφωνούν όλοι και έτσι θα, θα κάνουμε την προσπάθεια να ψηφίσουμε. Οι συντονιστές έχουν δώσει οδηγίες, μπορεί να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δεν είμαστε τόσοι πολλοί, δύσκολα χωνεύεται φαίνεται. Οπότε τελειώνει η ψηφοφορία. 17 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Η 201, όχι, η 524 ήταν. Η 184, ο εισηγητής είναι υπέρ, θέλετε να λάβετε το λόγο. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 184. Τώρα υπάρχει η 4160 Χάρτονγκ που κατεψηφίζεται. Η 525. Ποιος είναι υπέρ. Οι συγητές είναι υπέρ. Αλλά διαφέρουν οι απόψεις οπότε ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Θα ψηφίζω ώσπου να μου το απαγορεύσετε, λέει ο πρόεδρος. Λίγη ψηφοφορία. 17 υπέρ, 19 κατά, απερίφθη. 185. Η συγκίτρια είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, είναι η οπισθοφυλακή η οποία υιοθετείται. Μετά στο European Refugee Fund έχουμε τροπολογία 41-60 χάρτων που απορρίπτεται. Η 527 αποσύρεται, το ΕΛΚ δηλαδή αποσύρει την 527, όχι βέβαια, οπότε ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά εφόσον επιμένει το ΕΛΚ. Είμαστε 38 ψηφίσαντε, οι τρεις φαίνεται απέθαναν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού φαγητού, λίγη ψηφοφορία, 17 υπέρ, 18 κατά. Άρα απορρίπτεται. Υπάρχει η 4185 ε, για να ε, ε, ε, με συγχωρείτε, 41-95 ε, για ε, τα βασανιστήρια κατά των γυναικών. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπέρ. Πέρασε. δεν καλύπτει όμως την 41-96. Ε, Αφού βασανίσαμε τις γυναίκες τώρα τις συμπεριλαμβάνουμε. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Με συγχωρείτε. Μάλλον λάθος μου λένε. Η εισηγήτρια δεν συμφωνεί. Πρόκειται για την 41-96. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. 91-96 του κυρίου Σούριαν η συγγήτρια είναι ε, ε, αντίθετη ξεκινά λίγη η ψηφοφορία 13 υπέρ 22 κατά έχει απορριφθεί Περνάμε τώρα στην επόμενη γραμμή, μια νέα τροπολογία, πάντοτε στο ίδιο θέμα των βασανιστήριων κατά των γυναικών, 41-91. Ε, η συγγήτρια είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Είναι, ε, υπερψηφίστηκε. Επόμενη γραμμή για την ε, ενσωμάτωση των ε, υπηκών τριών χωρών. Ψηφίζουμε την 186. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η επόμενη καλύπτεται. Στην επόμενη γραμμή υπάρχει μία κλασική τροπολογία χάρτων που θεωρούμε ότι απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει και για τον επόμενο τίτλο 3 για το European Asylum Support Office. Και ε, κάτω στη σελίδα έχουμε μία τροπολογία ε, για τα ε, πιλωτικά προγράμματα, οπότε προχωράμε στη σελίδα 111. Έχουμε μία τροπολογία Ehrenhauser, κλασική. Όχι. Α, με συγχωρείτε. Είναι αποθεματοποίηση. Ποιος είναι υπέρ. Κανείς. Απορρίπτεται. Επίσης ε, αποθεματοποίηση του κυρίου Ερενχάουζερ, ε, οπότε υποθέτω θα ισχύει στο ίδιο. Η ε, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Υπάρχει προφορική τροπολογία της ε, εισηγητρίας. Πώς θέλετε να ψηφίσουμε, πέστε μου. <coughs> Θα ήθελα πρώτα να ψηφίσουμε την αρχική τροπολογία 702 702 που θα ήθελα να υπερψηφίσουμε. Αν καταψηφιστεί, προτείνω τροπο, προφο, τροποποίηση προφορική 1 εκατομμύριο 35. Και αν και αυτό καταψηφιστεί, 1.80. Ευχαριστώ. 702, tel qu'il est présenté là. Ε, ξεκινάμε λοιπόν από αυτή την τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Η συγκίτρια συμφωνεί κατά αποχές μία αποχή άρα υιοθετείτε. και όλες οι άλλες καταπίπτουν και του κυρίου Σούριαν όχι οπότε επανερχόμαστε στα βασανιστήρια η 41-93 ο είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ κατά όπως και πριν υπάρχει μία μικρή θετική ε, πλειοψηφία. 41-94. Η συγγήτρια είναι ε, υπέρ. Θα δεν υπάρχει ίδια πλειοψηφία, οπότε ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν δεν έχετε αντίρρηση, λέει ο πρόεδρος, θα ψηφίσω και εγώ. Λίγη ψηφοφορία, 17 υπέρ, 17 κατά, 2 αποχές, άρα απορρίπτεται. Κάτω στη σελίδα υπάρχει μια πιλωτική ενέργεια, γυρίζω σελίδα, όλη η επόμενη σελίδα είναι πιλωτικά προγράμματα. Φτάνω μέχρι το, γραφείο, το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Γραφείο European Police Office όπου υπάρχει σχόλιο του, της εισηγήτριας Europol Τι θέλετε να ψηφίσουμε Ήδη το είχαμε στον κατάλογό μας, στον κατάλογο ψηφοφορίας. So, all is done. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν έχουν καλυφθεί μέχρι και ε, ζητώ επιβεβαίωση από τον εισηγητή και την κυρία Χάου ε, το 4483 στο κάτω μέρος της σελίδας ε, έχετε μία πρόταση η κυρία εισηγήτρια μια οριζόντια για τις υπηρεσίες να αποκατασταθεί προσχέδιο η προφορική μου τροποποίηση είναι να το θέσουμε αυξημένο όμω το ποσό στο αποθεματικό. Υπενθυμίζω την αντίρρηση της Γιούτα σε μία άλλη πρόταση. Δηλαδή, αν έχει οθετηθεί σε κάποιο πακέτο, δεν μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τη συζήτηση για το πακέτο. Νομίζω μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό, διότι αν αποκαταστήσουμε το προσχέδιο, αλλά δεν έχουμε ψηφίσει τα σχόλια, δεν έχουμε ψηφίσει για την έρευνα όσον αφορά τις υπηρεσίες. cet amendement n'était pas compris dans l'accord général sur les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 ε, ή περιλαμβάνεται ή στη συζήτηση για, και την ψηφοφορία για τις οργανώσεις. Προφανώς όχι, άρα μπορούμε να το ψηφίσουμε. Ναι, αλλά έχουμε, ε, έχω σημειώσει ότι έχουμε συμφωνήσει για τη Europol. Εδώ είναι το Police College, δεν είναι η Europol. Οπότε, είναι προφορική τροπολογία, δηλαδή όχι αυτά που γράφτηκαν και πώς θα θέλετε να βάλετε στο απόθεμα. Θα ήθελα 425.000 να εγγραφούν στο αποθεματικό. Donc, ça veut dire que le chiffre qui... Δηλαδή, ο αριθμός ο οποίος είναι εδώ θα ε, πάει με πλάγια γράμματα και ε, για απόθεμα, ο σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξέρουμε τους όρους για την απελευθέρωση του αποθεματικού. Τι βρίσκεται ως λόγος πίσω από αυτή τη δημιουργία του αποθεματικού για την απελευθέρωση του. Δεν το έχουμε δει γραπτός, γι' αυτό ρωτάω. Το ερώτημα είναι σωστό. Τι απαντάτε. Εφόσον η κυρία Χάουγκ η Ακαδημία, η Αστυνομική Ακαδημία έχει μάλλον ένα πιο πρόβλημα και το λέω αυτό ανοιχτά και ειλικρινά. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα. Είχαμε πει ότι εδώ Όλα αυτά αποκαθιστούν το προσχέδιο προϋπολογισμού 425.000 ευρώ. Εντάξει. Και αν και όταν η Σιδόνια θέλει να το εγγράψουμε αυτό στο αποθεματικό, αυτό συσχετίζεται κάπως με την, πώς να το πω, πώς λέγεται, με την χορήγηση απαλλαγής που αυτή τη στιγμή υπάρχει τροχοπέδηση υποθέτω. Η δική μου τροπολογία λέει αποκατάσταση προσχεδίου προϋπολογισμού σε σχέση με το ποσό ναι, ακριβώς. Η Επιτροπή Ελέγχου προπολογισμού, η Επιτροπή Ελέγχου θα προτείνει την Ευρωπόλ για το έτος 2008 να μην χορηγήσουμε απαλλαγή. Α, συγγνώμη, Ακαδημία της ΕΠΟΛ, να μην χορηγήσουμε στην ΕΠΟΛ ε, Χωρί απαλλαγή. Να μην τις δώσουμε την απαλλαγή για την εκτέλεση του προπολογισμού. Συμφωνώ απόλυτα να πούμε αυτά τα 525 λέει η ομιλήτρια τώρα θα εγγραφούν στο αποθεματικό και ως όρο έχουμε ότι όλες οι προϋποθέσεις του όρου που έχουν θέσει ως όρο οι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού θα πρέπει να επιτευχθούν. Αυτό είναι όλο και όλο αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι λογικό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κατάλαβα. Καταρχήν δεν έχουμε ήδη ψηφίσει αυτή την τροπολογία, άρα μπορούμε να την ψηφίσουμε. Δεύτερον, ότι ε, προέρχεται η τροπολογία αυτή από τον, ε, την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού για να δίνει απαλλαγή σε κάποιο οργανισμό. Τι πιστεύει η, η συγγήτρια, θέλει το λόγο η Αν. Η Αν επειδή ουσιαστικά δεν λέει κάποιο όρο η προϋπόθεση εδώ, δεν τον δίνει. Είναι πολύ σημαντικό να είναι σαφής η όρη και οι προϋποθέσεις για την απελευθέρωση. Λείπει νομίζω αυτό, δεν βρίσκεται σε αυτήν την τροπολογία της Γιούτα. Τα Ναι, η δική μου τροπολογία ούτω ή άλλω είναι να αποκαταστήσουμε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προπολογισμό. Η συντόνια θέλει όμως αυτή η τροπολογία προφορικά να τροποποιηθεί και πάλι. Και μάλιστα να αποκαταστήσουμε το σχέδιο ναι μεν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όμως το ποσό να εγγραφεί στο αποθεματικό. Και ο όρος για την απελευθέρωση του αποθεματικού θα είναι ότι η ΣΕΠΟΛ, η ΣΕΠΟΛ θα υλοποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και άμεσα κιόλα στο προσεχές μέλλον, που δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι όροι και αυτές οι προϋποθέσεις ακόμα. Εγώ τουλάχιστον δεν τους γνωρίζω. Η κυρία Όλμαϊερ, παρακαλώ. Το πρόβλημα είναι ότι στην ΣΕΠΟΛ Έχουμε σοβαρές παρατυπίες και εδώ και χρόνια δεν έχουν αποσαφινιστεί και δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό τον λόγο από πλευρά συναδέλφου Ματιέ έχει εξεταστεί σε βάθος από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και κατέληξαν στο αποτέλεσμα για να πιέσουν την Επιτροπή επιτέλους να θέσει σε τάξη τα πράγματα επειδή έχουν πολλά κονδύλια εξαφανιστεί, πολλά χρήματα έχουν φτάσει σε χέρια ιδιωτών τα μοιράστηκαν κάποιοι. Για να υπάρξει λοιπόν πίεση, να αποκατασταθούν τα πράγματα και να αποκατασταθεί η τάξη, υπάρχει αυτός ο όρος. Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο περιορισμός τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ουσιαστικά το σχόλιο αποβλέπει στο να πούμε ότι το ποσό αυτό τοποθετείται στο απόθεμα μέχρι ότου εξεταστεί η κατάσταση αυτή της οργάνωσης από την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Με τέτοιο λοιπόν σχόλιο και με τέτοια παρουσίαση η συγγήτρια συμφωνεί ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή, άρα υιοθετείται προφορική τροπολογία. Ο κύριος Φαν, μπορούμε να ζητήσουμε από την εισηγήτρια να υποβάλει κάτι γραπτό ως πρόταση προτού καταλήξουμε στην Ολομέλεια μετά από την ψήφιση εδώ, γιατί αυτό θα ήταν χρήσιμο. Tout à fait légitime, Πολύ σωστό και γυρίζω σελίδα. Είμαστε πάντοτε στο European Police College. Υπάρχει μία τροπολογία 4160 που θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Η επόμενη γραμμή είναι η 526. Ποιος είναι υπέρ? Ηλεκτρονικά. Γιατί πιστεύω ότι... Ε, θα είναι τσίμα τσίμα. Είμαστε στην 526. Ε, Λίγη η ψηφοφορία. 20 υπέρ 19 κατά και ε, εγκρίνεται η τροπολογία. Η 43-60 αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία προφορική τροπολογία. Έχω μια προφορική τροποποίηση εδώ για μια υφιστάμενη τροπολογία που κατατάθηκε από τον κύριο Άλβαρο συζητήθηκε σε τεχνικό επίπεδο θα σας το διαβάσω το κείμενο τι λέει το αρχικό κείμενο λέει με ιδιαίτερη έμφαση τονίζει το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Η προφορική τροποποίηση λέει προδιαγραφές σε συγκεκριμένα θέματα συμπεριλαμβανομένης και της κυβερνοασφάλειας. Ευχαριστώ. If it is as it stays... Αν είναι όπως αναφέρεται και έχει συνταχθεί από το συντάκτη, δεν μπορώ να το υποστηρίξω, διότι θεωρώ ότι αλλάζει η νομική βάση. Αν δεχτείτε όμως την προφορική τροποποίησή μου, μπορώ να το δεχτώ. Cet amendement oral vous convient. Vous auriez à ce moment-là le soutien du rapporteur, et peut-être de son groupe. Maybe because I haven't seen the... Ίσως επειδή δεν είδα την συμφωνία που έγινε σε τεχνικό επίπεδο, θα μπορούσα να συμφωνήσω να πούμε ειδικά, ιδιαίτερα, αντί να πούμε συμπεριλαμβανομένη της, να πούμε ιδιαίτερα της, especially, αντί including. Λοιπόν, κατόπιν αυτού υποβάλλω την τροπολογία 4360 σε ψηφοφορία όσοι έχει συνταχθεί. Θέλετε πρώτα να ψηφίσουμε την τροπολογία, ναι, πριν τελειώσει, ε, γιατί είναι, προφορική. Ε, ε, πιστεύω το περιεχόμενο είναι λανθασμένο, αλλά θα τη δεχτώ. Λοιπόν, προφορική τροπολογία του εισηγητή με αποκαρδιωμένη αποδοχή από τον ετούντα την τροπολογία, ε, την 4360. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, 509 καταπολέμηση του εγκλήματος. Η ΣΥ είναι αντίθετη συγγήτρια εναντί αυτής της τροπολογίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, αλλά απορρίπτεται η τροπολογία. 65, cybercrime του κυρίου Αλβάρο. Υπέρ, κατά. Ε, από το η πράσινη είναι αντίθετη. Αποχές εγκρίνεται. Ε, το τέλος της σελίδας και η αρχή της επομένης καλύπτονται, πρόκειται για οργανισμούς. Και στο 46-56 έχουμε μία τροπολογία Ερενχάουζερ και ψηφίζουμε μετά τη 206. Η, η συγγήτρια είναι υπέρ την πρόληψη της, ε, των ναρκωτικών. Εγκρίνεται. Περνάμε στο Prince. Πρόκειται για τον τραγουδιστή, τον Prince. Υπάρχει η τροπολογία 843. Η, η συγκίτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Βλέπω ότι ο τραγουδιστής έχει ορισμένους ε, υποστηρικτές αλλά πολλούς ενάντιους και απορρίπτεται. 202 προτείνεται από την συγκίτρια. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4361 του κυρίου Άλβαρο. Η συγγήτρια είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Γυρίζω σελίδα. Είμαι στην 116. Επάνω. 203 της Επιτροπής Ελευθεριών, η συγκήτρια είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 203 και τελειώσαμε με το 3α. Και περνάμε στο 3β. Πιλωτικά αύριο. Κύριε Νάουζερ, Ναζέρα. υποκατηγορία, την 4688 ψηφίσουμε υπέρ. Κανεί κατά, καταπίπτει. Το ίδιο θα ισχύσει για τις παρόμοιες τροπολογίες του κυρίου Αρχάζη για αυτή την κατηγορία, 282. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. πιλωτικά προγράμματα μετά. Culture Program 4307 χωριστή ψηφοφορία το ποσό και τα σχόλια. Για το ποσό η συγκέντρια είναι κατά υπέρ, κατά <laughs> και ο συντάξης τροπολογίας είναι κατά αποχές, μασοχιστικές τάσεις εδώ μέσα. Ο, ο, συντάκτης απέριψε το ποσό και η, και η Επιτροπή το απέριψε. Τα σχόλια, ο εισηγητής είναι υπέρ των σχολείων. Η εισηγήτρια, συγγνώμη. Κα, κατά αποχές, πλειοψηφία, να δεχτούμε τα σχόλια. Δεν έχουμε λεφτά, αλλά λέμε τι, πώς θα χρησιμοποιηθούν. 3.14. υπέρ, 314 υπέρ, κατά, οι πράσινοι ούτε να απέχουν δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Κουλτούρα, ε, πολιτισμός, εκπαίδευση δεν τους ενδιαφέρει τους πράσινους. 6-10. Εδώ είναι οι γλώσσες που διατρέχουν κίνδυνο. Πέρα. Συγητής είναι εναντίον. Ποιοι είναι υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Le vote est Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ακόμα ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. 30 υπέρ. 8 εναντίον, μία αποχή διασφαλίσαμε, εξασφαλίσαμε και προστατεύουμε τις ε, απειλούμενες γλώσσες 43-31 καλύπτεται πρέπει να ψηφίζουμε την 573 η συγκιτρια είναι εναντίον ποιοι είναι υπέρ κατά οι φιλελεύθεροι δεν έχουν άποψη είναι υπέρ σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία c'est Και πρόκειται εδώ για την διεθνική κυκλοφορία και εμπορία πολιτιστικών προϊόντων. Τέλος ψηφοφορίας 20 υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε. Οι τροπολογίες στο κάτω-κάτω της σελίδας καλύπτονται και το ίδιο ισχύει και για την 118 με την εξαίρεση της ε, τροπολογίας αυτής που είναι στάνταρ τροπολογία και απορρίπτεται η χάρτον τροπολογία. Τώρα, ετήσια ειδικά γεγονότα και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια ειδική τροπολογία στη 43 γήτρια. Έχω μια προφορική τροποποίηση πράγματι για την 4303. Να αλλάξουμε το ποσό δηλαδή από 9 εκατομμύρια σε 4 εκατομμύρια και σε υποχρεώσεις και σε πληρωμές. Και δεν έχω άλλη κάποια τροπολογία για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις. Μπορούν να μείνουν όσοι έχουν. Η σύστασή μου είναι να υπεψηφιστούν. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι η ίδια τροπολογία με την τροπολογία του ΕΛΚ? 551. Όχι. Τι διαφορά έχει. Τα σχόλια. Όταν είδα την τροπολογία 4303 και την τροπολογία 551 του ΕΛΚ, η τροπολογία του ΕΛΚ δεν προσθέτει τίποτα, πιστεύω εγώ, στην πρώτη τροπολογία. Αν η 4303 εγκρίθει, τότε εγώ πιστεύω ότι η 551 καταπίπτει. καταπίπτει. Bon. James Ellis, Κύριε James Ellis. Έχουμε νούμερο ότι δεν μπορούμε να βάλουμε ποσό όταν είναι το earmarking. Εδώ τι γίνεται με τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, γιατί πάμε να ορίσουμε ποσό. Σωστή παρατήρηση αυτή του James Ellis. Η απάντηση είναι ότι αυτή τη γραμμή θα την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά από ό,τι τις άλλες, όντως. Σουριάν. Ο κύριος Σούριαν, δεν θέλω να αναλώσω τον χρόνο σας υπερβολικά, αλλά αν έχω δίκιο, πιστεύω ότι όταν έχουμε μεγάλο καλάθι, και προκαθορίσουμε και πούμε δύο εκατομμύρια από αυτό το καλάθι θα πάνε για αυτό και τον άλλο σκοπό. Αυτό είναι προκαθορισμός, earmarking. Αν έχετε όμως ε, μια, ένα κονδύλιο ξεχωριστό, δεν είναι earmarking, είναι ένα κονδύλιο με συγκεκριμένο ποσό που το πρικοδοτεί. Συγγνώμη, χάνουμε πέντε εκατομμύρια, αλλά εντάξει, έστω, αυτή είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Ε, η κυρία Εισηγήτρια, πρόεδρε, να υπενθυμίσω αυτό που είπα στην αρχή της συνεδρίασής μας σήμερα το πρωί, ότι υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που έχουν αυτό το πρόβλημα που θέτουν. Αναφέρουν ένα ποσό, το οποίο προφανώς δεν είναι ορθό, δεν είναι σωστό. Αυτό που είπα λοιπόν το πρωί ήταν ότι αυτή η φράση θα πρέπει πάντα, πάντα να αντικαθίσταται από ένα τμήμα που θα λέει ότι θα καλύπτεται μέρος των ε, υποχρεώσεων, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι λιγότερο χιδαίο λοιπόν ε, να πούμε, από το να πούμε marking. κύριε Σφάν, για αυτό το θέμα πιστεύω ότι το λογικό πράγμα να κάνουμε θα ήταν να διαγραφεί όλο αυτό το κονδύλιο. Δεν το προτείνω να το κάνουμε, αλλά στο μέλλον να το δούμε αυτό, διότι αν έχουμε ένα κονδύλιο ετήσια έκτακτα γεγονότα ή εκδηλώσεις, είναι αδύνατο να αποφύγει κανείς το earmarking. Τι μπορεί να κάνει κανείς. Ετήσια γεγονότα και εκδηλώσεις είναι, πρέπει να αναφέρονται και κάτι να πάρουν. Το earmarking είναι αναπόφευκτο, αναπόφευκτη συνέπεια του να υπάρχει ένα τέτοιο κονδύλιο που εντάσσουμε. Ίσως θα συμφωνήσουμε του χρόνου να διαγράψουμε απόλυτα αυτή τη γραμμή. Πολύ ωραία, δεν τολμούσα να την πω, αλλά όντως πρέπει να έχουμε μία γραμμή κατά επεισόδιο. Special annual events, τέτοιες εκδηλώσεις, εκατομμύρια. Αυτά για του χρόνου, το πάντων, για τις εκδηλώσεις του χρόνου. Προς το παρόν σας προτείνω να ψηφίζετε αυτή την προφορική τροπολογία με το νέο νούμερο, 4 εκατομμύρια, που προτείνει η Συντόνια 4303, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Καλύπτονται οι δύο επόμενες. Δεν καλύπτει το ομως όμως 42-91. Ψηφίζουμε. Et rapporteur est contre. Oui. Le rapporteur est contre. Qui est pour Η συγκέντρια είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 41-64 του κυρίου Μοργκάντη. Εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 43-06 Γκάγερ. Εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Ο κύριος Γκάγερ είναι υπέρ αυτή τη φορά. Κατά. Αποχές. Λυπάμαι κύριε Γκάγερ, απορρίφθηκε. 41-64 Μοργκάντι και οι άλλοι και γυρίζουμε σελίδα. 273 Επιτροπή Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά προπαρασκευαστικές δράσεις σελίδα 121. Μέχρι το Deutsch Stammes, 4168. Κυρία Συγγήτρια, τι θα κάνουμε. Είχαμε ψηφίσει για το ποσό στην οριζόντια τροπολογία όμως θα έπρεπε να ψηφίσουμε τις παρατηρήσεις, οι δύο τελευταίες τροπολογίες σε αυτή, σε αυτή τη γραμμή. Ευχαριστώ. Μόνο τα σχόλια. Τη 4168 εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μεγάλη πλειοψηφία. Απομονωμένο το έργο εδώ. 42-02 το ίδιο. Μόνο τα σχόλια. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι επόμενες τροπολογίες είναι πειραματικά προγράμματα και μία του Χάουζερ που απορρίπτεται. Όχι, όχι, έχουμε μία Χάουζερ 4681. Ω, 10% είναι και αυτή. Πάει και αυτή. Europe for Citizens Expenditure καλύφθηκε. Multimedia Actions. Η συγγήτρια θα μας προτείνει να ψηφίσουμε πρώτα την 625 με προφορική τροπολογία της Αν Γένσεν, η οποία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό που συνέβη είναι ότι ήρθαν σε επαφή μαζί μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας ότι δεν τους αρέσει πολύ αυτή η τροπολογία η 625. Αν την αποσύρουμε, είπαν, αυτό που θα έκαναν θα ήταν να δεχτούν, θα δεχόντουσαν να έχουμε μια τροπολογία που θα ζητούσε ένα στρατηγικό σχέδιο, στρατηγικό προγραμματισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τα κονδύλια για τις πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που είχε ζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου επί μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αυτό που προτείνω τώρα λοιπόν είναι ότι έχουμε μια ευκαιρία μπροστά μας τώρα, ένα παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται για να έχουμε ένα ποσό στο αποθεματικό και όρο για την απελευθέρωση του αποθεματικού ότι θα δοθεί αυτό το στρατηγικό σχέδιο προγραμματισμού για την Επιτροπή Πολιτισμού ώστε να γνωρίζουμε πώς αυτά τα χρήματα θα δαπανηθούν στο μέλλον όταν θα αυξήσουμε τα ποσά για την πολιτική ενημέρωσης και πληροφόρησης. Πιστεύω είναι μια καλή λύση αυτή. <clears throat> αν υπάρξει υποστήριξη για αυτό το αίτημα εδώ και νομίζω ότι η κυρία Γεντρογεύσκα έχει τη σωστή διατύπωση για αυτή την τροπολογία, ε, τότε θα πρότεινα να αποσύρουμε την τροπολογία που έχουμε καταθέσει, την 625, για τις παρατηρήσεις. Και θα αφορούν τώρα τις δαπάνες για περισσότερους ε, δημοσιογράφους, φωτογράφους και τα που περιτριγυρίζουν τον κύριο Μπαρόζο. Αντί να πούμε δεν θέλουμε να, κάνει, να γίνεται αυτό, λέμε δώστε μας ένα στρατηγικό προγραμματισμό για την πολιτική πληροφόρηση και ενημέρωσης. Είναι ένας πιο θετικός τρόπος στη διατύπωση. Καταλαβαίνει τον πολιτικό στόχο Σαλβαντόρα. Δεν έχω τίποτα εναντίον τέτοιων προτάσεων και τροπολογιών και όρους και προϋποθέσεις για το αποθεματικό. Το ερώτημα είναι πώς και πού θα συζητηθεί αυτό το στρατηγικό πρόγραμμα και σχεδιασμός. Διότι δεν νομίζω ότι είναι της Επιτροπής Προϋπολογισμών, αλλά είναι θέμα διαθεσμικής ομάδας επικοινωνίας ή κάποιου τέτοιου φορέα. Είναι οι σωστές προϋποθέσεις και όροι που πρέπει να εξειδικεύουν περισσότερο τους όρους για την απελευθέρωση. Πώς δέχεται δηλαδή η Επιτροπή Προϋπολογισμών μια τέτοια προσέγγιση. Θα ήθελα να μας δοθεί μεγαλύτερη αποσαφήνιση ποιοι θα είναι οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν αν αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός, το στρατηγικό αυτό πρόγραμμα θα γίνεται δεκτό ή όχι από μας. Ευχαριστώ ο κύριος Φάρ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι υποτίθεται ότι πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 277 της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων. Δεύτερον, είμαστε κατά του αποθεματικού. Είχαμε προγράμματα επιπρογραμμάτων, στρατηγικά έγγραφα για την ενημέρωση και πληροφόρηση. Δεν νομίζω να επαναληφθεί και να είναι χρήσιμο να επαναλαμβάνεται αυτό. Ευχαριστώ. Ελγα Τρούπερ, υποστηρίζω πάρα πολύ την προσέγγιση της συναδέρφου για αυτή την τροπολογία. Ξέρετε ότι εργάζομαι στην Επιτροπή Πολιτισμού και έχω παρακολουθήσει όλες τις συζητήσεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας και τι μας υποσχέθηκαν και ότι θα μας έδιναν μέχρι τώρα. Πρέπει να δοθεί ένα μέσο, ένα εργαλείο για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό υποστηρίζω το αίτημα της συναδέλφου. Κύριος Μπέγκε παρακαλώ. ο περισσότερο προσωπικά να συμφωνήσω με τον Γιώραν Φάρμ Πιστεύω και εγώ ότι η πολιτική ενημέρωση και πληροφόρηση είναι το συγκεκριμένο προνόμιο και δικαίωμα κάθε ενό θεσμικού οργάνου. Κάθε ενό θεσμικού οργάνου. Και γι' αυτό η Επιτροπή Προπολισμών έχει δικαίωμα να ζητήσει να μάθει τι γίνεται με τα κονδύλια αλλά σε σχέση με τη γενική γραμμή για την πολιτική και πληροφόρηση θα πρέπει να είμαστε κάπω πιο επιφυλακτικοί. Τώρα αυτό που διοργανικά συμφωνείται διαθεσμικά με πολύ κριτικό πνεύμα πρέπει να εξετάζεται στη συνέχεια και εκεί το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να διεξαγάγει μια σε βάθος συζήτηση γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται καμιά φορά η εντύπωση ότι αυτά που είναι κέντρα βάρους για την ενημέρωση πληροφόρηση για το επόμενο έτος μέσα από τη διοργανική συμφωνία από την Επιτροπή χειραγωγούνται και εμείς τρέχουμε πίσω από αυτό για να δούμε τι έχει γίνει και το κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι σειράκι οποιοδήποτε. Πρέπει να παρακολουθεί, να βλέπει τι γίνεται. Αλλά αλλού στο Προεδρείο και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ίσω πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Χρειάζεται μια διαφορετική συζήτηση από ό,τι αυτή που έγινε στο παρελθόν για να επιληθεί το πρόβλημα. Κύριο Άλβαρο παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και για την προθυμία της να λάβει υπόψη αυτές τις προτάσεις και να τις εξετάσει θετικά. Ταυτόχρονα για τον συνάδελφο Φέρμ και κύριο Μπέγκε για αυτά τα οποία πρότεινε η κυρία Τρούπερ, το είπε η Άννε Γένσεν, είχε η Επιτροπή Πολιτισμού ζητήσει επί πολλά χρόνια να υπάρξει ένας προγραμματισμός αυτών των θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά τα χρήματα είναι ένα τμήμα των 20 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δώσει πιο ευδιάκριτο ρόλο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω φωτογράφων που θα είναι διαθέσιμοι επί 24 ώρες για αυτόν ε, τηλεοπτικών συνεργείων. Αυτό δεν είναι όμως στρατηγική για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Είναι απλά και μόνο η παρουσία πολλών ε, δημοσιογράφων ε, που θα παρακολουθούν τον πρόεδρο. Τώρα, Τώρα, για να κάνουμε κάτι για να διευκολυνθεί η Επιτροπή, δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτά τα κονδύλια τα οποία δεν τα αμφισβητούμε, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν αν θα υπάρξει και αύξηση αυτών των 20 εκατομμυρίων. Να, να πούμε αν είμαστε πρόθυμοι να δούμε, να δώσουμε αυτά τα κονδύλια, πείτε μας εσείς πώς θέλετε να δώσετε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω, πώς θα πετύχετε καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση. Και είναι συμφέρον μας ε, και το Ευρω... ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και εμάς τους ίδιους μας αφορά αυτό το θέμα της επικοινωνίας και εμένα και άλλους συναδέφους που πρέπει να εκθέσουμε στις εκλογικές μας περιφέρειες αυτά τα οποία γίνονται και δεν, δεν ε, μπορούμε να υπομισθούμε τις ευθύνες γενικών διευθυντών. Η κυρία Άννα Γένσελ παρακαλώ έχει τον λόγο. Απλά και μόνο για να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσε ο Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Νομίζω ότι η αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Πολιτισμού. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Επιτροπή Πολιτισμού να πάρει ένα εργαλείο, ένα μέσο στα χέρια της που δεν είχε μέχρι σήμερα για να κάνει τη δουλειά της. Πρέπει να υποστηρίξουμε θα λέγα, αυτό το αίτημα και προς τον Ράιμερ Μπέργκε και την κριτική που άσκησε θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αρχική τροπολογία της ομάδας Άντε είναι το να ξεκινήσει αυτό και αυτά άλλαξαν απόλυτα με την προφορική τροποποίηση που υπέβαλε η εισηγήτρια διότι με αυτήν ανατράπηκαν τα πράγματα, γύρισαν τα πάνω κάτω. Όχι για την ανάμειξη πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα, αλλά λέμε εξηγήστε τι θα γίνει στον τομέα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Είναι κάτι που η Επιτροπή Πολιτισμού προσπαθεί εδώ και πολύ καιρό και έχει καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, ότι αυτό πρέπει να γίνει, γιατί είναι πρόβλημα πώς επικοινωνούμε πώς περνάει το έργο που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα έξω και πώς διοργανικά και διαθεσμικά μπορεί να προχωρήσει προς τα έξω ώστε να είναι κατανοητή και ε, εύκολα κατανοητή η Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πολίτες. Και σε σχέση με αυτά τα σχέδια, προγράμματα, σχέδια, για να προσελκυστούν οι πολίτες στην Ευρώπη, δεν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Θέλουμε οι πολίτες να έχουν ευκαιρία να καταλαβαίνουν τι διάολο γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το σημαντικότερο είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια σωστή διατύπωση τώρα που θα είναι θετική, θα στρέφεται προς το μέλλον και θα υποστηρίζεται και από την κυρία Ρέντινγκ γιατί λέει ότι θα τηρήσει την υπόσχεσή της. Αλλά να έχουμε ένα μέσο, ένα εργαλείο στα χέρια μας, να την κάνουμε να τηρήσει τα υπεσχημένα, αυτά τα οποία δεσμεύτηκε να κάνει ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Όλοι έχετε το γραπτό κείμενο της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Να στο το διαβάσω. Το ποθ... Μπαίνει στο αποθυματικό. Το ποσό, το ποσό μπαίνει στο αποθυματικό μέχρι ότι η Κομισιόν παρουσιάσει μια συνολική στρατηγική με στόχο το πώς τα όργανα της Ένωσης θα επικοινωνούν καλύτερα με τον Ευρωπαίο πολίτη με βάση την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου Κομισιόν με τίτλο «Επικοινωνία με εταιρική σχέση στην Ευρώπη» από τον Οκτώβριο 2008. Ψηφίζουμε αυτή την προφορική τροπολογία 625 η συγγήτρια θέλει το λόγο. Η συγγήτρια είμαι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Νομίζω σωστά εξισορροπεί τις άλλες τροπολογίες. Πρέπει εδώ να πούμε σαφώς ποιο θα είναι το ποσό το οποίο θα εγγραφεί στο αποθεματικό. 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Και η ταπεινή μου πρόταση πώς θα έπρεπε να ψηφίσουμε, νομίζω από κοινού με την τροπολογία 277 θα έπρεπε να την ψηφίσουμε αυτή την πρόταση. Διότι αποκαθιστάτε έτσι, αποκαθιστάτε με συγχωρείτε το προσχέδιο προϋπολογισμού. Και έτσι και με αυτό το οποίο είχαμε πει με την προφορική τροποποίηση, με την επιχειρηματολογία που μόλις μας διαβάσατε. Ευχαριστώ. Oui, ce même. On vote d'abord les chiffres. Ωραία, πρώτα ψηφίσουμε το πόσο το ποσό. Μετά θα δούμε το αποθηματικό. Τώρα το, το ποσό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε το ποσό. Τώρα το αποθεματικό. τι συνθήκες να βγει από το αποθεματικό υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό εγκρίθηκε. αγγελίθηκε. 43-51 αποσύρεται. Τελειώσει με τα multimedia. Σελίδα 123. Κλασική Ερενχάουζερ. 207. Εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Κανένας. Ο κύριος Βόπος, μόνο ένας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι φιλελεύθεροι αποσύρουν την 6 προς 6. 43-52 καλύφθηκε. Information outlets. Μία Ρενχάουσερ κλασική. 308 Επιτροπή Πολιτισμού, Το κονδύλιο για τις δυνατότητες πληροφόρησης ενημέρωσης μετά από τις διαπραγματεύσεις μας. Προτείνω ένα χαμηλότερο ποσό να εγγραφεί προφορική τροποποίηση για 980.000 και στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές 980.000 αντί 1,5 εκατομμύρια ευρώ. 980.000. au groupe socialiste. Et Τίνεται προ του σοσιαλιστέ που τη δέχονται. Λοιπόν, προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε. Και αυτό καλύπτει τι δύο επόμενε. Ρενχάουζερ κλασική. Επόμενη σελίδα 124, 840. Εισηγήτρια κατά. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 41-49. Αρτών κλασική. 4630 46-30. Ερχάους καλύπτεται. 208 Υπέρ, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι. Κατά. Οι περισσότεροι, τα μαμούθ είναι κατά. Τα μαμούθ συντρίβουν αυτή την τροπολογία. Public Opinion Analysis. Κλασική χαρτών. Απορρίπτεται. 46-16 Ερενχάουζερ επίσης. 2.78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46-35 Ερενχάουζερ κλασική 209 Europe for Citizens υπέρ κατά ο μεγάλος στρατός κατά απορρίπτεται 4189 κλασική χαρτόγκ απορρίπτεται οι δύο άλλες στη σελίδα 125 είναι προπαρασκευαστικές δράσεις 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τριακόσα δέκα. Εισηγήτρια υπέρ. Όχι, κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 603 πιλωτικό γυρίζουμε σελίδα 4670 κλασική Ερεχάζερ και 4676 552 ΕΛΚ υπέρ ηλεκτρονικά η 552 Αποσύρεται. Η επόμενη είναι 553. Το ΕΛΚ μπορεί να αποσύρει αν θέλει. Όλοι θα χαρούμε. Και την αποσύρει το ΕΛΚ. Μπορεί ένα σύστημα. Αν αποσυρθούν όλες οι τροπολογίες ΕΛΚ και σοσιαλιστός, είναι ένας καλός τρόπος να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Αρτών 554. Αποσύρεται. Εξαιρετικό αυτό. 253. Υπέρ. Πολύ. Κατά. Τρεις. Αποχές εγκρίνεται. 403 καλύφθηκε. Σχόλια του 430. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέλος της European Food Safety Authority. Καλύπτεται από τις υπηρεσίες. 128. 41-61 η υπόλοιπη σελίδα, πιλωτικά προγράμματα. Θα πάμε στο Civil Protection Within the EU. το 668 των σοσιαλιστών. Που την αποσύρουν. Τι λέω Γκέρα, να αποσύρει. Αποσύρθηκε, ωραία. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα της 4304. Πρέπει να την ψηφίσουμε. 4304. Υπέρ. Κανένας. Απορρίπτεται. 395. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γυρίζω σελίδα. Κατηγορία 4. Και σταματάω. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, όλα τα μέλη, τους συνεργάτες. Τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο το πρωί στις 9 να μείνουν οι συντονιστές και η Έλγα κυρίως η Έλγα Τρία λεπτά διακοπή.